Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Ξαναρχίζουμε τις εργασίες μας. Ε, τα πρακτικά της χθεσινής ημέρας διανεμήθηκαν. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει από αυτόν. Ως εκ τούτου εγκρίνονται τα πρακτικά.